Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξή μας. Πρώτα απ' όλα όμως να κάνω και μια ανακοίνωση, ε, μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου με πρόταση για απόφαση η οποία ε, είχε υποβληθεί χθε, είχε περιθώριο 24 ωρών και επομένως βάσει του άρθρου 6 τη δεχόμαστε την πρόταση αυτή ως έχει. Αύριο στην 20 η Μαΐου του 2015 ε, θα αναφερθεί ως μεταξύ των εγγράφων που θα πρέπει να μοιραστούν. Συνεχίζουμε. Κοινή συζήτηση για την νομιμοποίηση εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ε, σύσταση για δεύτερη